So, colleagues, we are going to, uh, to start again. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ας περάσουμε στις ψηφοφορίες. Καθίστε παρακαλώ. Il n'y a que des votes électroniques, hein, on est d'accord oui. okay. I'm going to chair in French. So... Στα γαλλικά θα προεδρεύσω, οπότε αν χρειάζεται, βάλτε τα ακουστικά σας. Λοιπόν, Ψηφίζουμε πρώτα την πρόταση για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Ακόμα και αν δεν ήθιστε, μια που υπάρχουν πολλοί νέοι εδώ και είναι κείμενα που τώρα ανακαλύπτουμε, θα πρότεινα να δώσουμε το λόγο ε, στον εισηγητή για ένα λεπτό για να μας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Ο Κρίστοφ Χάνσεν λοιπόν που είναι η συγητής της Επιτροπής μας για αυτό το πρώτο κείμενο και για να μας εξηγήσει. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πράγματι, πρόκειται για να διατύπωση της οδηγίας για το πόσιμο είδωρ. Κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια ουσιαστικά. Πρόκειται για την ε, πρωτοβουλία πολιτών που έχει συγκεντρώσει 1,5 εκατομμύριο υπογραφές για να υπάρχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό, αλλά και για την ποιότητα του ύδατος, του πόσιμου, αλλά και για ό,τι έρχεται σε επαφή με το νερό αυτό. Έτσι λοιπόν, έχουμε κοιτάξει με τους κοιόδες εισηγητές ποια είναι τα βασικά στοιχεία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι είναι αυτό που πρέπει να υποστηρίξουμε απέναντι στο Συμβούλιο, μια που δεν βρισκόμαστε στην ίδια γραμμή. Ο Μισελ Νταντάν στην προηγούμενη θητεία είχε στα χέρια του αυτό το φάκελο. Ε, ψηφίσαμε στην Ολομέλεια. Τώρα πρόκειται απλώς για την εντολή προκειμένου να μπούμε σε διαπραγματεύσει σε τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ψηφίζουμε λοιπόν με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα τις ψηφοφορίες. Ωραία, μπράβο. Καλά δουλέψατε. Έχουμε μια ευρία πλειοψηφία προκειμένου να μπούμε σε τριμερή διάλογο. Περνάμε τώρα στην δεύτερη ψηφοφορία που αφορά την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. Λίγο πολύ το ίδιο θέμα που μας ε, επιτρέπει να μπούμε σε τριμερή διάλογο. Θα δώσω το... Α, δεν είναι εδώ κυρία Σίμωνα Μποναφέ από ό,τι βλέπω. Οπότε θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα της ψηφοφορίας. Καλώς. Οπότε θα αρχίσουν οι τριμερείς διάλογοι που αρχίζουν έτσι κι την επόμενη εβδομάδα για αυτά τα δύο θέματα. Εύχομαι ε, πολύ δύναμη στους διαπραγματευτές μας. Περνάμε στην τρίτη ψηφοφορία τώρα. Είναι ψηφοφορία για την προφορική ερώτηση που έχει να κάνει με το COP25. Θα μιλήσουμε δηλαδή μετά σήμερα αργότερα, εδώ δεν, δεν ψηφίζουμε το ψήφισμα, αλλά την προφορική ερώτηση, έτσι, που θέτει η Επιτροπή μας. Πρώτη ψηφοφορία για την προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. δεύτερη ψηφοφορία για το ίδιο θέμα, αλλά για το Συμβούλιο. Ψηφίστε. Πέρα της ψηφοφορίας. Και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία των όσων συζητήσαμε σήμερα το πρωί. Πρόκειται καταρχήν για την αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράταση των περιόδων έγκρισης ε, διάφορων ε, δραστικών ουσιών ε, μεταξύ άλλων της φυσικαμίνης και άλλων. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η αντίρρηση. Απλή πλειοψηφία χρειάζεται. Περνάμε στη δεύτερη ψηφοφορία, για τη δεύτερη δηλαδή αντίρρηση. Πρόκειται για την παράταση των περίοδων έγκριση δραστικών ουσιών διάφορων ε, ουσιών, μεταξύ άλλων του κλωροτολουρών. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Υπάρχει πλειοψηφία για την αντίρρηση. Συνεχίζουμε και περνάμε σε τρεις ψηφοφορίες για τρεις ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Είναι αντίρρηση για τη διάθεση στην αγορά διάφορων προϊόντων και ξεκινάμε με το MZHG0JG. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η αντίρρηση. Δεύτερη πρόκειται για την τροποποιημένη σόγια Α274 του 12. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Και περνάμε εδώ στην επόμενη ψηφοφορία για διάφορους γενικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Υπάρχει αντίρρηση λοιπόν και για τα φυτοφάρμακα και για τους γενετικά τροποποιημένους αυτούς οργανισμούς. Πέρας των ψηφοφοριών. we are going to... Λοιπόν, συνεχίζουμε και περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή COP25 στη Χιλή. Έχουμε ένα ψήφισμα το οποίο έχει υπογραφεί από έξι πολιτικές ομάδες και θα δώσω το λόγο στις έξι αυτές πολιτικές ομάδες και αρχίζουμε με το ΕΛΚΑ και τον Πίτερ Λίζε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Ε, έχω εμπνευστεί από το πάθος εκατομμυρίων ε, νέων ανθρώπων οι οποίοι ε, έκαναν ό,τι μπορούσαν στους δρόμους για να εισακουστούν οι φωνές τους. Ε, μπορεί αυτό, αυτό να το είπε ένας πράσινος πολιτικός, αλλά δεν ήταν αυτός που πράγματι το είπε, ήταν η εκλεγήσα απρόεδρος, η νέα πρόεδρος της Επιτροπής, η Ursula von der η οποία πραγματικά ε, θεωρεί πως έχει εμπνευστεί από αυτήν την ε, από το πάθος ε, των νέων για την προστασία μας από την κλιματική αλλαγή και νομίζω πως ε, όλοι μας θα πρέπει να εμπνευστούμε με ίδιο τρόπο από τους νέους μας και ότι θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη δική μας πλευρά προκειμένου να αυξήσουμε την προστασία μας από την κλιματική αλλαγή και να κάνουμε να προβούμε σε συγκεκριμένα μέτρα για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τις αεροπορικές μεταφορές μεταφορές και άλλου τομεί του οποίου δεν έχουμε κάνει αρκετά μέχρι στιγμή, Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές ε, έχουμε συζητήσει επανειλημμένα αυτό το ζήτημα μεταξύ των συντονιστών ε, και θεωρούμε πραγματικά κάτι το εξαιρετικά δυσάρεστο, το, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναφέρει ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν αλλά ταυτόχρονα η αντίστοιχη οργάνωση από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, συνεχίσει με το σύστημα εμπορίας εκπομπών στον αερο, ε, αεροπορικό τομέα και νομίζω πως στις δύο διασκέψεις που θα λάβουν χώρα, ειδικότερα στο Μοντρεάλ, στο εγγύς μέλλον, θα πρέπει να το κάνουμε αυτό γνωστό και να επιστήσουμε την προσοχή του κοινού σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να υποστηρίξουμε την προσέγγιση της ε, Προέδρου Ποντελάιν και επίσης ε, θα πρέπει να κάνουμε και αυτό που προσέθεσε ότι δηλαδή θα πρέπει εδώ να μην αναλάβουμε δράση μόνοι μας, θα πρέπει να το κάνουμε από κοινού με τους πολίτες μας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ε, δεν θα υπάρξει και κατάλληλη υποστήριξη ε, δεν μπορούμε δηλαδή έτσι απλά να αποφασίσουμε κάτι πολύ γρήγορα εδώ. Όχι, θα πρέπει να ενθουσιάσουμε τον κόσμο και να πείσουμε του πολίτε, ειδικότερα για παράδειγμα του ανθρώπου που δουλεύουν στον τομέα ε, τον, ε, του άνθρακα ε, ή αλλού, έτσι ώστε να θελήσουν και εκείνοι να κάνουμε αυτή την δίκαια μετάβαση. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν αντιδράσει μέσα στα επόμενα χρόνια. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι το γεγονό ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο και οι νόμοι τη φυσική επιβάλλουν αυτή την πραγματικότητα του ότι μπορούμε εμεί να κάνουμε ό,τι θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών και ούτω καθεξή, αλλά ταυτόχρονα είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαζόμαστε με τρίτες χώρε για να επιτύχουμε ε, κάτι περισσότερο. Δηλαδή, Ασκούνται συνέχεια κριτικέ εδώ σε εμά και στι εθνικέ κυβερνήσει ότι δεν κάνουν αρκετά, αλλά στα διάφορα φόρα των Ηνωμένων Εθνών διαπιστώνουμε ότι τελικά είμαστε οι μονόφθολμοι, οι οποίοι δηλαδή βασιλεύουμε ανάμεσα στου τυφλού. Οπότε ε, ας το έχουμε και αυτό κατά νου όταν θα κάνουμε τι προτάσει μα σε ό,τι αφορά αυτή την πρόταση ψηφίσματος μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από σοσιαλιστές, Ευχαριστώ. Από τους σοσιαλιστές ο, Μωαμέντε Να δω, δουλεύει το μικρόφωνο μου. Δουλεύει. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε χρόνο μιλίας. Και αυτό μου τι να πω. Ε, εδώ στην Επιτροπή μας για την ΚΟΠ. Ειδικά αυτές τις δύο εβδομάδες όπου νέοι ακτιβιστές για το κλίμα διαδηλώνουν και ζητούν να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή. Μας ζητούν να είμαστε πιο τορμηροί. Τους στόχους πρέπει να δούμε, τις φιλοδοξίες που έχουμε ως Ευρώπη και πώς μπορούμε να εμπνεύσουμε και τον υπόλοιπο κόσμο για να είναι λιγάκι πιο ουδέτερος απέναντι στο κλίμα τουλάχιστον. Η συνεισφορά μου λοιπόν δεν θέλω να στραφεί προς το πώς θα γίνουμε πιο τολμηροί και πιο φιλόδοξοι στους στόχους. Το θέμα είναι πώς θα γίνει μια δίκαιη μετάβαση. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη κάνουν αυτό που υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν. Είναι δύο πολύ σημαντικά πράγματα αυτά για τους σοσιαλιστές στην Ευρώπη. Σοσιαλδημοκράτες και σοσιαλιστές στην Ευρώπη. Θα μπορούσα να πω πολλά για το κλίμα, την κλιματική δικαιοσύνη, όπως και το ΕΛΚ. Και εμείς περιμένουμε τα σχέδια της Κομισιόν. Από τα πρώτα που είδαμε μπορούμε να πούμε ότι είμαστε θετικά διακείμενοι. Έχουμε ένα ειδικό ταμείο για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να γίνουν πιο κλιματικά ουδέτεροι και να έχουμε και καλύτερου στόχου. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για τη δικαιοσύνη και την εφαρμογή. Πού έχουμε φτάσει, ούτω ώστε όταν πάμε στη Χιλή να παίξουμε ηγετικό ρόλο για να γίνει καλύτερο ο πλανήτη μας. Θα πρέπει να πούμε σε αυτούς τους νέους που διαδηλώνουν αυτές τις εβδομάδες ότι τους ακούμε και ότι κινούμαστε κι εμείς προς σωστή κατεύθυνση. Θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες από την ομάδα μου, ε, ώστε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Αυτά, δεν, δεν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο. Ευχαριστώ. Από το Renew, Νίλς Τόρβαλτ. Ε, Πριν από έξι εβδομάδες είχα μια ειδική σύνοδο στην Εύη με την Επίτροπο. Η... Κατά την ομιλία της ε, υπήρχε μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Σχεδόν έκλαψε χθες στον ΟΗΕ. Αλλά σχεδόν είχε κλάψει και τότε όταν μας ε, είχε μιλήσει εδώ στην Επιτροπή μας. Είχε μια πολύ συναισθηματική προσέγγιση λοιπόν. Και το ίδιο συνέστημα το βλέπουμε και σε εκατοντάδες χιλιάδες νέων. Μερικές φορές ε, τα συναισθήματα είναι καλά, εξυπηρετούν πολιτικούς σκοπούς. Αλλά μερικές φορές ελοχεύουν και κινδύνους, για, ειδικά όταν είναι περίπλοκα τα θέματα. Άκουσα λοιπόν τους νέους, όπως η Γκρέτα Τούμπερ, και θυμάμαι όταν ήμουν νέος εγώ, όταν μιλούσαμε για τις τρίτες χώρες, και ίσως σκητούσαμε με ένα βλέμμα που ε, έδειχνε ότι δεν καταλαβαίναμε όλες τις ε, πτυχές του τρίτου κόσμου. είναι δύσκολο να καταλάβουμε τις περιπλοκότητες αυτών των θεμάτων. Αν δείτε την ε, έκθεση για την περιβαλλοντική αναθεώρηση της, κομιδιών, της Κομισιόν που δημοσιεύτηκε φέτος, θα καταλάβετε τι σας λέω. Αυτές οι εκθέσεις δείχνουν ότι κάποιες χώρες όπως και η δική μου, η Σουηδία, τα πάνε καλά σε ό,τι αφορά την πορεία που έχουν ακολουθήσει για να υλοποιήσουν του στόχου. Αλλά υπάρχουν πολλέ άλλε ευρωπαϊκέ χώρε που δεν είναι σε τόσο καλή θέση όσο οι δικέ μα χώρε. Γι' αυτό θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι όταν προσπαθούμε να βρούμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για το πρόβλημα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και τι ε, διαφορέ των χωρών. Το πόσο διαφορετικέ είναι οι ευρωπαϊκέ χώρε. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα επιτύχουμε στι προσπάθειές μας και για αυτό που είπαν οι σοσιαλιστές για την δίκη μετάβαση. θα τα καταφέρουμε. Είναι περίπλοκο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Μερικές φορές έχουμε την αίσθηση ότι θα γίνει καλύτερος ο κόσμος ε, αν χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρίες. Αλλά και με, ας πούμε, δεν θέλουμε όμως να καίμε τα τροπικά δάση στο Κονγκό για να πάρουμε αυτά τα μέταλλα και να φτιάξουμε τις μπαταρίες. Δεν το θέλουμε αυτό. Είναι περίπλοκο το θέμα και θα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλες τις λεπτομέρειες, ε, όλα τα περίπλοκα προβλήματα ας πούμε, που είναι συνειφασμένα με αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Πράσινη. Παρ Χόλγκρεν. Δεν είναι εδώ. Γιάννη Ευχαριστώ. Όταν ήμασταν στο Κατοβίτσε, πριν από ένα χρόνο σχεδόν, ήταν το μεγάλο ραντεβού που δικαιολόγησε την αποτυχία του Κατοβίτσε. ήταν η σύνοδος του ΟΗΕ και όλοι λέγανε ότι ναι, δεν τα καταφέραμε στο Κατοβίτσα, θα τα καταφέρουμε στη σύνοδο του ΟΗΕ. Θα είναι έτοιμη η Ευρώπη, θα γίνουν νέε δεσμεύσει, θα δείξουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να δώσουμε το παράδειγμα και όχι μόνο να διδάσκουμε από καθέδρα. Όταν βλέπουμε την ε, έκθεση η οποία ε, εκδόθηκε σήμερα το πρωί, δεν είναι το θέμα ότι είμαστε λιγότερο κακοί. Το θέμα δεν είναι να είμαστε λιγότερο κακοί από του άλλου. Δεν μπορούμε να είμαστε αυτάρισκα και να λέμε, αφού έχουμε τη Βραζιλία, τι Ηνωμένε Πολιτείε, τη Ρωσία, η Ευρώπη τελικά ε, πάει και άσχημα. Όχι. Πάει άσχημα. Επί χρόνια η ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό αφήγημα ήταν ότι εμεί είμαστε καλύτεροι από του άλλου. Άρα μια χαρά είμαστε. Μην κρίνετε την Ευρώπη, μην την επικρίνετε, μια και είναι και καλύτερη από του άλλου. Αλλά η δική μα δουλειά ω ευρωβουλευτέ, δεν είναι να είμαστε καλύτεροι από του άλλου. Είναι να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, που οφείλει να κάνει και να δώσει το παράδειγμα σε όλο τον πλανήτη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε μέχρι τη Χιλή, με αυτή τη νέα κομισιόν στο πλευρό μας, είναι να πείσουμε με το παράδειγμά μας. Όχι μόνο να είμαστε δραστήριοι, να είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, στην ΚΟΠ, αλλά να πείσουμε με το παράδειγμά μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τους στόχους μας σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου μέχρι το 2030 Υπάρχει μια συζήτηση, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διεκδικήσει το ότι ο ευρωπαϊκός στόχος σε ό,τι αφορά το κλίμα δεν είναι ένα στόχος που αποφασίζεται στη Σύνοδο Κορυφής, αλλά με συναπόφαση. Εξού και η συζήτηση που κάνουμε για το, την νομοθεσία για το κλίμα. Και να αυξήσουμε τους στόχους μας, να αυξήσουμε τις, δεσμε, τις ε, επενδύσεις ό,τι αφορά τα κτίρια, τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις μεταφορές. Επομένω, πρέπει να κάνουμε το μάθημά μα για να δώσουμε το παράδειγμα. Δίνοντα το παράδειγμα, σημαίνει ότι δείχνουμε και αλληλεγγύη απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο, κυρίω απέναντι στι χώρε που δυσκολεύονται. Τι ξέρουμε αυτέ τι χώρε, που είναι τα πρώτα θύματα τη απορρίθμιση του κλίματο και είναι και λιγότερο υπεύθυνε παρόλα αυτά. Α δείξουμε λοιπόν, α ας δώσουμε το παράδειγμα τι κάνουμε για να μεταβούμε σε μια άλλη κατάσταση Ας δούμε ε, την έκθεση που εκδόθηκε σήμερα με το, για τον 1,5 βαθμό και ας είμαστε ε, αλληλέγγυα απέναντι στις άλλες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τι έχουν ε, υποφέρει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η συνάντηση αυτή του κόπο στη Χιλή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι όπως ήταν στο Παρίσι, όπου καταλήξαμε σε μια συμφωνία ή όπως ήταν στο Κατοβίτσε. Τώρα βλέπουμε τους νέους να κατεβαίνουν στο δρόμο και να ζητούν περισσότερες δράσεις. Αν δείτε τις αποφάσεις του Παρισιού, θα δείτε ότι ήδη αυτές είναι πολύ δύσκολο να τεθούν σε εφαρμογή και η Κατοβίτση συνάντησε και έδειξε ακριβώς αυτή τη δυσκολία. Παρά ε, τις επιτυχίες που είχαμε, επειδή μία χώρα λέει όχι, δεν καταλήξαμε σε συμφωνία. Σήμερα λοιπόν το πιο σημαντικό θα ήταν να διασφαλίσουμε ότι ό,τι συμφωνήθηκε στο Παρίσι και οτιδήποτε συμφωνήθηκε στο Κατοβίτσε να υλοποιηθεί όσο γίνεται καλύτερα και παντού ανά τον κόσμο πέρα από το ότι υπέγραψα και εγώ το ψήφισμα για το COP25, να ξέρετε ότι είμαι κατά μονομερών αλλαγών στους στόχους του 2013 από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς πρέπει να περιμένουμε και πρέπει να περιμένουμε ε, τι θα κάνουν και άλλοι του 2030 βέβαια. Ναι. Πρέπει να περιμένουμε γιατί αλλιώ αν ε, περιμένουμε τους άλλους ε, δεν θα γίνει τίποτα. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο να διασφαλιστεί η ισορροπία ανάμεσα στις εκπομπές και ε, τις μειώσεις ε, που θέλουμε για το 2050. Τώρα κάποιες χώρες, σε κάποιες περιοχές όπως και στην Πολωνία θα έχουν τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος από τέτοια μέτρα. Υπάρχει ενεργειακή ένδυα σε μας και σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε ακόμα κανένα άλλο σχέδιο B. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιαν το ανέφερε. Είπε, αναφέρθηκε στην μετάβαση την ενεργειακή, ε, κάτι το οποίο μας δημιουργεί κάποιες ελπίδες, αλλά ίσως εσείς δεν αντιλαμβάνεστε το κόστος το οποίο θα κληθούμε να επομιστούμε στην Πολωνία. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, πάντως ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με θή τρόπο. Η Πολωνία ήδη αποφάσισε την ε, ηλεκτρική κινητικότητα. Είναι κάτι που έχει μεγάλη σημασία σαν θέμα. Επίσης μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και για την αποψήλωση των δασών. Έχουμε πολλά καλά παραδείγματα και έχουμε πολλούς φιλόδοξους στόχους για περισσότερα δάση, 33% μέχρι το 2050. Επίσης αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πράγματα στις πόλεις. Το σχέδιο προσαρμογής που ετοίμασε η Πολωνία ε, ήταν ε, κάτι που κρίθηκε πολύ θετικό και ικανοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτά ναι, αλλά να μην αναλάβουμε δράσεις οι οποίες βραχυπρόθεσμα μεν θα μας δοξάσουν, αλλά μακροπρόθεσμα θα μας επιφέρουν ζημιά. Τελευταίος, ο μιλητής για τον ε, πρώτο γύρο, Wallace. Εκ μέρους της Γκουε. Η ορθολογική εταιρεία πριν από μερικούς μήνες έστειλε το μήνυμα ότι αυτά που κάνουμε όχι απλώς δεν φτάνουν, αλλά είναι μάλλον και άχρηστα αν δεν κλείσουμε το χάσμα μέχρι το 2030, δεν θα πετύχουμε τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Πρέπει να αυξήσουμε τις φιλοδοξίες μας, αν θέλουμε να περιοριστεί η θέρμανση του πλανήτη κάτω από τον 1,5 βαθμό. Ο πρόεδρος Τάσκα αυτή την εβδομάδα εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πόσο καλά τα καταφέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επίπεδο της κλιματικής φιλοδοξίας όμως της Ευρώπης δεν συνάδει με τη Συμφωνία των Παρισίων. Όχι, δεν κάνουμε ό,τι πρέπει στην Ευρώπη. Το ψήφισμα μας έλεγε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα για να μειώσουμε μέχρι το 2030 κατά 25% τις εκπομπές σε σχέση με τη δεκαετία του 90. Ε, το ψήφισμα που έχουμε μπροστά μας δεν αναφέρει καν ποσότητα, καν ένα ποσοστό. Θέλουμε να κάνουμε μια τροποποίηση τι, για να περιορίσουμε τις φιλοδοξίες των Παρισίων. Το σχέδιο ψηφίσματος που έχουμε μπροστά μας πάντως θα πρέπει να το ξαναδούμε. Έχουν γίνει πολλά και έχουν αλλάξει πολλά τα τελευταία χρόνια. Το διακυβερνητικό πάνελ για το κλίμα τα λέει και τα ξαναλέει ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγές στην οικονομία μας. που δεν ελήφθη υπόψη καν στα συμπεράσματα της διάσκεψης 24. Ε, πολλά ήδη απειλούνται με εξαφάνιση. Είχαμε τον πιο ζεστό Ιούλιο ποτέ. Εμείς λοιπόν θέλουμε το ψήφισμα αυτό να λέει κάποια πράγματα με νόημα, να έχει νόημα. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να κάθεται και να παριστάνει τον τροπαλό. Εμείς εκπροσωπούμε τον κόσμο κανονικά. Τον κόσμο που κατεβαίνει στους δρόμους σε τέτοια νούμερα, 4 εκατομμύρια το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και θα έχουμε ακόμα περισσότερου. Δεν μπορούμε λοιπόν να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και να βλέπουμε του νέου μόνο σε κινητοποίηση. Ευχαριστούμε. Ξεκινάει τώρα η διαδικασία Catch the Eye, στο πλαίσιο τη οποία κάθε μέλο ε, μπορεί να πάρει το λόγο για 1,5 λεπτό. Οπότε μην διστάσετε να σηκώσετε τα χέρια σας θέλετε να πάρετε το λόγο. Δυνατότητα λοιπόν από το ΕΛΚ, παρακαλώ ως πρώτη ομιλήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή μας ε, για ε, τη δουλειά που έχει γίνει σε σχέση με αυτό το πολύ σημαντικό ψήφισμα ε, και νομίζω πως όλοι μας συμφωνούμε πως ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής είναι εξαιρετικά σημαντικός και σε κάθε περίπτωση έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον αγώνα. Τα κράτη-μέλη είναι βέβαια υπεύθυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 9% των παγκοσμίων εκπομπών και γι' αυτό ε, στην δική μου ε, κατά τη δική μου άποψη, σε αυτό το κείμενο του ψηφίσματο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μόνη τη τι προκλήσει που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει δηλαδή να αναλάβουν την ε, απαραίτητη δέσμευση όλε οι χώρε προκειμένου να έχουμε αποτελέσματα. Και κατά τη δική μου άποψη, θα πρέπει οι στόχοι μα ε, σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή να επιτευχθούν με τρόπο που να μην υπονομεύσουν την ανταγωνιστικότητά μα, χωρί δηλαδή να ωφεληθούν από αυτό άλλες τρίτες οικονομίες. Η Κίνα, για παράδειγμα, υπενθυμίζω ότι είναι ήδη υπεύθυνη για το 25% των παγκοσμίων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ενώ αναμένεται πως θα αυξήσει περαιτέρω έως το 2030 τις εκπομπές της. Άρα λοιπόν θεωρώ πως είναι απαραίτητη η ανάληψη παγκόσμιας δράσης για να καταπολεμήσουμε επιτυχώς την κλιματική αλλαγή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ για την συμμετοχή αυτή. Υπάρχουν πολιτικές δεσμεύσεις, η Κίνα, η Ινδία, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ένα, μια πολιτική δέσμευση πολύ χαμηλότερη από αυτό που θα θέλαμε οι πιο νέες γενιές δίνουν μάθημα στον κόσμο, όμως δεν μπορούμε μόνο με δεσμεύσεις, μόνο με λόγια ε, να λέμε ότι συμφωνούμε. Πρέπει να σταθούμε στο ύψος των ευθυνών μας και να αναλάβουμε υποχρεώσεις, πραγματικές υποχρεώσεις που συνδέονται με την φορολογία. Αυτός είναι ο δρόμος. Οι κυρώσεις επίσης για τους κλάδους της γεωργίας, της ενέργειας ή των μεταφορών. Αν δηλαδή δεν προσθέσουμε υποχρεώσεις με δίκαια φορολογία ή με ένα καθεστώς κυρώσεων στα επίπεδα του στόχου που θέλουμε να πετύχουμε θα είμαστε αδύναμοι. Ενώ δεν πρέπει να είμαστε αδύναμοι, πρέπει να είμαστε ισχυροί. Τώρα ήρθε η ώρα να περάσουμε σε δράσεις και να αναλάβουμε υποχρεώσεις. Δεν έχουμε κανέναν για το Renew, οπότε περνάμε στους ε, πράσινους, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπε ο προηγούμενος συνάδελφος, ότι δηλαδή ενδεχομένως δεν θα πρέπει ε, να είμαστε πολύ συναισθηματικοί σε σχέση με την ανάληψη αυτή τη Είδαμε 4 εκατομμύρια ανθρώπου όμω στου δρόμου το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Ένα 4 εκατομμύρια ανθρώπου μόνο στη Γερμανία. Οπότε λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο κίνημα το οποίο έχει δημιουργηθεί και καλά θα κάνουμε εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβουμε σοβαρά υπόψη μα αυτό το κίνημα. Γιατί πραγματικά θα πρέπει εδώ να γίνουν αλλαγέ. Θα πάμε λοιπόν για μία ακόμα φορά ε, στη Χιλή χωρί να αυξήσουμε τη δική μα ε, ε, δέσμευση. Οπότε αυτό καταδεικνύει στου πολίτε μα ότι δεν μα ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα και δεν είναι καλό αυτό στο πλαίσιο μια δημοκρατία δεν νομίζω ε, πω η συνάδελφοι μας λέει ότι δεν θα πρέπει να είμαστε πολύ συναισθηματικοί. Ουσιαστικά διαβάζει αυτό που αναφέρει η έκθεση του IPCC. Και τι αναφέρεται μέσα σε αυτή την έκθεση. Γιατί τι αναφέρεται εκεί, ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο, γιατί σε καμία περίπτωση ε, ε, θα οδηγηθούμε σε μία ε, κατάσταση θερμοκηπιακή όπου θα αυξάνεται συνέχεια η θερμοκρασία και θα φτάσουμε στους 46, ε, κατά 46 βαθμούς ε, πιο υψηλή θερμοκρασία, ένα περιβάλλον δηλαδή στο οποίο δεν μπορεί να επιβιώσει ο άνθρωπος. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ ε, αντικειμενικά δεδομένα και δεν είναι τίποτα συναισθηματικό. Διαβάζοντα αυτό το ψήφισμα, ε, μου γεννιούνται διάφορα ερωτηματικά για την ε, ορθότητα αυτών των συστάσεων. Καταρχάς, οικονομικά. Πώ θα ξεκινήσουμε το 2020 και θα έχουμε σταθερή οικονομικέ συνεισφορέ να γνωρίζουμε τι ε, δυσκολίε των βορείων χωρών να κινητοποιήσουν τέτοια ποσά. Επίση, ε, τι εγγύσει έχουμε ότι αυτό το ταμείο θα το διαχειρίσουν, θα το σωστά οι δικαιούχοι. Ε, υπάρχουν και άλλα σημεία προβληματικά. Από τη μία, η ατζέντα που έχουν βάλει ε, οι ειδικοί των ε, ΜΚΟ που μιλούν για παγκόσμια δράση, ενώ η απάντηση βρίσκεται στην τοπική και εθνική συνεργασία από την άλλη μια κλιματική φιλοδοξία μη ρεαλιστική, ενώ ξέρουμε ότι οι στόχοι του Παρισιού δεν θα υλοποιηθούν. Αρκεί να δούμε τον πραπτασιασμό των εργοστασίων που χρησιμοποιούν άνθρακα ε, στην Ασία και τις, την αποψήλωση των δασών και τις πυρκαγιές στην Αφρική και στην Λατινική Αμερική. Επίσης χρησιμοποιείται η κλιματική διπλωματία ε, για να υποσκάψει την εθνική κυριαρχία των κρατών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σοσιαλιστές. Αλεξάνδρα Μορέτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους εισηγητές. Θαυμάσια δουλειά τους. Η COP25 θα είναι μια κρίσιμη στιγμή για να υλοποιήσουμε αυτά που αποφασίσαμε στο Παρίσι. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία και δεν πρέπει να τη χάσουμε. Θα πρέπει να είμαστε στο ύψο των προσδοκιών των νέων που κατέβηκαν σε διαδηλώσει και αυτέ τι μέρε σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο στοιχεία που κατ' εμέ πρέπει να τα εμβαθύνουμε περισσότερο. Καταρχά το θέμα τη υγεία και το άλλο το θέμα των γυναικών. Για το θέμα τη υγεία. Με, με βάση μια πρόσφατη μελέτη του, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία ανάμεσα στο 30 και το 50 θα έχουμε 250.000 θανάτους το χρόνο λόγω κακής διατροφής, ελονοσίας και ε, θερμοπληξίας. Κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή θα έχει, όπως όλοι ξέρουμε, μια επίπτωση όλο και μεγαλύτερη στα εθνικά συστήματα της υγείας, με κοινωνικό κόστος όλο και υψηλότερο. Αυτό δεν θα επηρεάσει μόνο την ε, υγεία των ασθενών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί θα παράσχουν βοήθεια και θα παίξουν το ρόλο τους και θα κάνουν τη δουλειά τους. Επομένως, θα υπάρχει σημαντική επίπτωση στη δημόσια υγεία. Θα αυξηθούν κάποιες αρρώστιες, π.χ. οι αλλεργίες. Η εγκυμοσύνη των γυναικών. Πολλές γυναίκες και πολλές μελέτες δείχνουν ότι θα υπάρχουν πολλές αρρώστιες ε, στις εγκύους... και πολλές, πολύ πρόωροι τοκετοί. Ε, θα έχουμε πολλά θνησιγενή έμβρια ε, παιδιά μάλλον, κάτι τη διάρκεια του τοκετού. Επίσης, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι γυναίκες αισθάνονται όλο και περισσότερο στο πετσί τους την κλιματική αλλαγή, πολύ περισσότερο από τους άντρες. Και αυτό γιατί δεν εμπλέκονται αρκετά στις ε, διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. Επομένως, θα πρέπει να δούμε και το θέμα του φύλου για, μελετώντας την επίπτωση της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τι επίπτωση θα έχει στο γυναικείο φύλλο η κλιματική αλλαγή. Όλος ιδιαίτερο. Ευχαριστούμε. Εκ μέρου των Πρασίνων, η κυρία Πάουλου. Ευχαριστώ. Θέλω να τονίσω ότι κάποιοι εδώ λένε ότι μόνο 9% έχουμε τις ε, από τις ε, παγκόσμιες εκπομπές, όταν έχουμε 6,5% του πληθυσμού. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να πω ότι είναι λάθος αυτά που λέτε, αλλά αν η Γκρέτα Τούμπεργκ μπορεί να αλλάξει την κατάσταση και παγκοσμίω μέσα σε ένα χρόνο να βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα. Αν μια χώρα, η Γερμανία, μπορεί να υιοθετήσει μια νομοθεσία η οποία λέει ότι πάνω από 90% αύξηση στο κόστος για τα φωτοβολταϊκά, τότε νομίζω ότι στην αγορά όπου τόσοι μηχανικοί ερευνητές κάνουν πολύ καλή δουλειά με υψηλά έσοδα, θα έπρεπε να είναι σε θέση να κάνουν τη διαφορά στην COP25. Bah, ça écoute. Thank you. Um, maybe also to... Ευχαριστώ. Να πω και εγώ κάτι για αυτά που ακούσαμε εδώ. Με εκπλήσουν κυρίω αυτά που λένε οι συνάδελφοι από το ΕΛΚ που λένε ότι είναι πολύ σημαντικό το κλίμα, αλλά κατά τα άλλα ακούω μανιάνα. Α τα αφήσουμε για μεθαύριο. Σημαντικό, αλλά να μην βιαζόμαστε κιόλα. Μα Πρέπει να συμμορφωθείτε και πρέπει να καταλάβετε ότι η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιούργησε κάποιες προσδοκίες. Δεν ξέρω αν τα έχετε παρακολουθήσει στην ε, Νέα Ορκή τι έγινε. Ο Τάσκ είπε για το πακέτο για το 2030. Ναι, αλλά αυτά είναι η ρητορική των τελευταίων πέντε ετών και είπε ότι έχουμε κλιματική ουδετερότητα, ίσως κάποια μέρα να κάνουμε μεγάλη πρόοδο. Αυτά είπε η Ευρώπη στη Νέα Υόρκη. Ενώ από την άλλη η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργεί τεράστιες προσδοκίες και αυτό μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη. Λοιπόν, πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητα και αυτό το λέμε και στην Επιτροπή, γιατί περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει τις μεταρρυθμίσεις για το κόπο, γιατί έχει τεράστιες επιπτώσεις στο κλίμα. Και όταν ε, έρθουν με κάποια νομοθεσία τις πρώτες 100 μέρες για την ε, ε, και νομοθεσία για το περιβάλλον και για το κλίμα, να μην πάμε πάλι πίσω στις συζητήσεις που κάναμε τα τελευταία πέντε χρόνια και να λάβουμε υπόψη μας και τις ενέργειες μεταφορές και τις θαλάσσιες. Αυτό θα επιδράσει, αυτό περιμένει ο κόσμος και επιτέλους το ΕΛΚΑ ελπίζω να συμφωνήσει με αυτούς τους στόχους επιτέλους. Ο Πίτερ Λίζε. Συγγνώμη που παρεμβαίνω. Αλλά είναι μπας ε, η νιωστή φορά που φτάνεις καθυστερημένος στη συνδρίαση και μάλλον δεν παρακολούθησες τι είπα στην αρχή. θα πρέπει να αναθωρήσεις αυτά που είπες. Είναι απαράδεκτο να έρχεσαι αργά και μετά να τα βάζεις και με τις μεγάλες ομάδες. Δεν μας άκουσες όλους, οπότε νομίζω ότι πρέπει να πάρεις πίσω αυτά που είπες. Πείτε. 30 δευτερόλεπτα. Ξέρεις περί νέων τεχνολογιών κάτι. Ωραία. Λοιπόν, μπορεί να παρακολουθήσει τι συνεδριάσει των κοινωνιστικών επιτροπών και από το κομπιούτερ σου. Θα σου το εξηγήσω κάποια μέρα. Είναι φανταστική αυτή η τεχνολογία. Και σίγουρα δεν ε, μιλούσες για το μείον 55, μιλούσες ε, για τις ενέργειες μεταφορές, ναι, πάντα το κάνεις αυτό, αλλά επιτέλους πρέπει να γίνουμε συγκεκριμένοι για το μείον 55% το 2030. Και αυτό έχει φύγει από το ψήφισμα ε, χάρη στο ΕΛΚ. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι. Αν είσαι υπέρ του μείον 55% πες το στο ψήφισμα. Είσαι υπέρ. Πρόεδρος, εκτός μικροφώνου παρέμβαση από τον κύριο Λίζε. Πρόεδρος, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση σίγουρα. Και θα την έχουμε όταν φτάσουμε στις τροπολογίες που θα ψηφίσουμε για το ψήφισμα αυτό. Και θα σας πω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα σε λίγο. Τώρα τελευταίος από τους σοσιαλιστές η Goodland. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και για αυτή την τελευταία συζήτηση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό πραγματικά να μιλήσουμε για την φιλοδοξία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω, πείτε, μπορεί να μην είσαι εσύ το μεγάλο εμπόδιο, αλλά η ομάδα σου σίγουρα εκφράζεται με δύο διαφορετικές προοπτικές. Και εγώ ανησυχώ να λέμε 50% για το 2030, ενώ όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε παραπάνω. Και δεν θα ήθελα να υπάρχουν αυτές οι δύο γραμμές που καθυστερούν τελικά την υλοποίηση και την πρόοδο. Εμείς ως ε, θεσμικό όργανο είμαστε πολύ σημαντικοί για τους νέους και για τους ακτιβιστές για το κλίμα. Σήμερα λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε ότι δεν θα καθυστερήσουμε περισσότερο και να μην αφήσουμε ε, την Επιτροπή να πιστεύει ότι μπορεί να πορεύεται με δύο διαφορετικά ποσοστά, το 5% και το 55%. Να πιέσεις και εσύ την Επιτροπή να μην καθυστερήσει τις φιλοδοξίες μας για το 2030. Και βεβαίως θέλω να πω ότι συμφωνώ με τις προτεραιότητες της ομάδας μας όπως τις εξέφρασε ο κ. Σέιμ νωρίτερα. Μάλιστα. Α, τώρα γίνεται ενδιαφέρον. Α, τώρα αρχίζει να γίνεται ενδιαφέρον. Θα κάνουμε και άλλες συζητήσεις για αυτό το θέμα. Όταν πριν ψηφίσουμε. Θα δώσω το λόγο στην Γενική Διεύθυνση Κλίμα από την Κομισιόν. Πέντε λεφτά το πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής για τις σημαντικές παρεμβάσεις, πολύ ζωντανές. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα-δύο θέματα που προέκυψαν στη σημερινή συζήτηση, αν μου επιτρέπετε. Να πω δύο λόγια για το επίπεδο φιλοδοξίας. Να ασχοληθώ με το IMO και το ICAO και για τη συναντρίαση ε, στο Σαντιάγκο της Χιλής αρχές Δεκεμβρίου. Από Ευρωπαϊκή Σκοπιάς έχουμε εφαρμόσει το στόχο μας ε, μείωση 40% μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Έχουμε μια πλήρη νομοθεσία ε, που τη θέσαμε πολύ πριν τις υπόλοιπες μεγάλες ε, οικονομίες. Ε, όλοι μιλήσατε, ή κάποιοι μιλήσατε για την ε, εφαρμογή. Είναι σημαντικό για την Κομισιόν, για το Κοινοβούλιο, για το Συμβούλιο να εξασφαλίσουμε ότι εφαρμόζεται πλήρω αυτή η νομοθεσία και όπω ξέρουν πολλοί, αν εφαρμοστεί ε, πλήρω, Μπορούμε να φτάσουμε και πέραν του 40%, μπορούμε να φτάσουμε και στο 45% μείωση στι εκπομπέ. Επίση, το συζητήσαμε διαμακρό με τα κράτη-μέλη, με του υπουργού ε, περιβάλλοντο, στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο στο Ελσίνκι. Γίνεται και τεχνική δουλειά για το πώ ε, θα γίνει η επικαιροποίηση στα, στους στόχους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν, πώς μπορούν να προσαρμοστούν στο πλαίσιο που υπάρχει. Οποιαδήποτε αλλαγή στους βασικούς στόχους θα πρέπει να περάσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αυτό συνδέεται και με τη νέα νομοθεσία που έχει ανακοινώσει η υποψήφια πρόεδρος ε, για το κλίμα, που θέλει και τεχνική και πολιτική προετοιμασία. Η νέα Κομισιόν όμως θα το υποβάλει και όχι η τρέχουσα Επιτροπή. Ας, ε, Ας περιμένουμε λιγάκι να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βεβαίω, ε, πρέπει να προοδεύσουμε και τη μακροπρόθεσμη, με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική που πρότεινε πριν από κάνα χρόνο η Κομισιόν και που την, και μίλησε για αυτή και στην Κατεβίτσε, αλλά και στην Νέα Υόρκη. Ε, τα περισσότερα κρατημέλη συμφώνησαν για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και μας βάζει σε μια τροχιά για μια ουδέτερη Ευρώπη ως προς τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2050. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να μιλήσουμε ε, για το ότι η Κομισιόν και η επόμενη ε, Πρόεδρος θέλει την υποστήριξη των μαζών με τους τοπικούς φορείς, με τον κλάδο, με τη βιομηχανία, με τα σχολεία, με τους πάντες. Και η ιδέα για μια δίκαιη μετάβαση είναι πολύ σημαντική για να μην αφήσουμε κανέναν στο, πλευρό, στο ξεχασμένο από όλη αυτή τη διαδικασία εν ώψη των στόχων του 2050. Να πω δύο λόγια για το Σαντιάγκο. Ε, χαιρόμαστε με αυτό το ψήφισμα, γιατί και οι διαπραγματευτές χάρη σε αυτό, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν μια καλή ιδέα για το πώς αντιδράσουν στις ε, επερχόμενες διαπραγματεύσεις. Ξέρουμε ότι έκανε πολλά το Κατοβίτσε, έθεσε τους κανόνες διαφάνειας για τις ε, κυβερνήσεις, κανόνες που είχαν ε, συμφωνηθεί στο Παρίσι. Υπάρχει όμως ένα εκρεμές θέμα, τμήμα 6, μέτρα αγοράς. Προτεραιότητα για μας αυτό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει αυτό και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν υποσκάπτουμε την ε, περιβαλλοντική ακαιρεότητα. Κάτι τέτοιο θα ήταν αποδεκτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε φιλοδοξία, δεν θέλουμε να υπάρχει διπλή καταμέτρηση σε καμία περίπτωση, γιατί αυτά ήταν βασικά θέματα για την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συμφωνία του Παρισιού. Επίσης, στο Σαντιάγκο θα μιλήσουμε για το μηχανισμό της Βαρσοβίας που δεν θα πρέπει να υποσκαφθεί και γίνονται κάποιες συζητήσεις για την ε, το οικοδόμηση μηχανικού και για το σχέδιο ε, για τον αληθή υπόψη η διάσταση του φύλου. Για τους ωκεανούς, σίγουρα θα κάνει παρέμβαση και θα ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρξει πρόοδος και σε αυτόν τον τομέα. Πολλοί ομιλητές μίλησαν για την αεροπορία και την αυσιπλοεία. Και εδώ, η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαρη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε πλήρως το κεκτημένο μας. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι το σημερινό επίπεδο κλιματικών φιλοδοξιών σε ό,τι αφορά το ETS δεν υποσκάπτεται και οτιδήποτε προκύψει από το ICAO δεν θα προδικάσει την αναθεώρηση του συστήματος εκπομπή εκπομπών, το λεγόμενο ETS. Επίσης, θα πρέπει να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Θέλω να έρθω σε συνεργασία με, το, με τον ΙΚΑΟ, ούτω ώστε να έχουμε μακροπρόθεσμους στόχους για το μέλλον. Στον IMO είμαστε πολύ δραστήριοι. Θέλουμε βραχυπρόθεσμα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν πριν το 2023. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το πετύχουμε αυτό. Ξέρετε ότι η επόμενη πρόεδρος ε, στις πολιτικές κατευθυντήρες γραμμές έχει μιλήσει για αυτά τα δύο θέματα και θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η δουλειά με τη νέα επιτροπή το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Κλείνουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση. Τα επόμενα βήματα να σας υπενθυμίσω. Η προθεσμία για τις τροπολογίες επί του ψηφίσματος είναι 2, η Δευτέρα Οκτωβρίου μέχρι τις 11 ε, το βράδυ. Έτσι. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΕΜΒ στις 6 ή 7 Νοεμβρίου και στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο. Δεύτερη Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Στις 11 το πρωί, συγγνώμη, το βράδυ. Θα είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουμε εδώ να πάρουμε επίσημη θέση για το κλίμα από τη στιγμή που εκλεγήκαμε. Και είναι ακρογωνιαίος λίθος της πράσινης, της πράσινης συμφωνίας. Αυτό το ψήφισμα θα είναι σημαντικό και πολιτικά. Είναι σημαντικό λοιπόν όλα τα μέλη να συμμετάσχουν στη συζήτηση και στην ε, συζήτηση για τις τροπολογίες. Και στην ψηφοφορία βεβαίως που θα γίνει τον Νοέμβριο. Πολύ ωραία. Άρα θα πάμε στο τελευταίο θέμα για σήμερα. Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με το δεύτερο σχέδιο δράσης για να καταπολεμήσουμε το παράνομο εμπόριο καπνού. Ε, το ζήτησαν οι συντονιστέ. Πρώτοι οι σοσιαλιστές μάλιστα. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Όλαφ για να ξεκινήσει την παρουσίαση για 10 λεπτά. Και εν συνεχεία, αν συμφωνεί η ομάδα των σοσιαλιστών, θα τους δώσω το λόγο για να εξηγήσουν το αίτημά τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την παρουσίαση των 10 λεπτών από την Όλαφ. Thank you, Chair. Good afternoon. My... Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Ονομάζομαι Γκέο Γουίπλινγκ ε, και είμαι επικεφαλής ε, μονάδας στην Όλαφ το Γραφείο δηλαδή Καταπολέμηση τη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε ό,τι αφορά το παράνομο εμπόριο καπνού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν την Επιτροπή σα ε, για την πρόσκληση ε, που λάβαμε για να σα εξηγήσουμε σήμερα εδώ τι ακριβώ συμβαίνει με το παράνομο εμπόριο καπνού και τι ακριβώ κάνουμε για να τα πολεμήσουμε. Καταρχήν θα ήθελα να σα εξηγήσω πώ εμεί εξετάζουμε το φαινόμενο του εμπορίου καπνού. Ε, σήμερα και από εκεί και μετά θα σας πω τι κάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τι προσπαθούμε να κάνουμε ως νέες δράσεις ε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το είδος παράνομου εμπορίου. Καταρχήν λοιπόν να σας πω ότι όλο αυτό το Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως εντολή τον εντοπισμό, την διερεύνηση και την πρόληψη της απάτης όταν αυτά τα φαινόμενα σχετίζονται με τα τα, και τα, τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης έχουμε εν, μια εντολή ακριβώς διερευνητική, ενώ έχουμε και μια εντολή πολιτικού χαρακτήρα. Τι είναι λοιπόν ε, το τόσο σημαντικό προκειμένου ακριβώς να αντιμετωπίσουμε το παραγωγικό εμπόριο καπνού. Ουσιαστικά υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι. Πρώτον, υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα τα οποία ε, είναι διαφυγόντα ε, και είναι χρήματα των φορολογούμενων αυτά. Γνωρίζετε δηλαδή πόσο υψηλή είναι η φόρη στα προϊόντα καπνού και ε, θεωρούμε πως ε, Εάν όλα αυτά τα προϊόντα λοιπόν είχαν υποβληθεί κανονικά σε φόρους, θα είχαμε εξοικονομήσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως των φορολογούμενων μας. Και επίσης βέβαια γνωρίζετε πόσο σημαντικές είναι οι πολιτικές υγείας οι οποίε διέπουν αυτά τα προϊόντα. Δηλαδή, οι τιμέ καθορίζονται ακριβώ στο λόγο των πολιτικών υγεία και το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού οδηγεί στο να υπονομεύονται αυτέ οι πολιτικέ. Τέλο, ένα τρίτο λόγο είναι το γεγονό ότι υπάρχουν ε, θέματα ασφαλεία που σχετίζονται με αυτό το είδο ε, παρανομού εμπορίου. Δηλαδή, πρόκειται για έναν κλάδο εντό εισαγωγικών στον οποίο δραστηριοποιούνται οι οργανωμένε εγκληματικέ οργανώσει με χαρά μου ε, έχω διαπιστώσει ότι η Όλαφ και κατά την προηγούμενη θητεία ε, το Κοινοβουλίου έλαβε ισχυρή εντολή προκειμένου να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά ε, αυτό το φαινόμενο και αναμένουμε με ενδιαφέρον την νέα σας θητεία από την πλευρά του Κοινοβουλίου προκειμένου να συνεχίσουμε αυτή την κοινή προσπάθεια. Να σας εξηγήσω τώρα τι ακριβώς κάνουν οι αρχές των κρατών μελών, οι συνοριοφύλακες, δηλαδή οι αστυνομικές αρχές ε, και όλες οι συναρμόδιες αρχές προκειμένου να απομακρύνουν αυτά τα προϊόντα από την αγορά. Βλέπουμε λοιπόν μια σταθερή τάση κατά τελευταία χρόνια όπου ε, έχουμε κατασχέσεις γύρω στα 3 ε, με 4 δισεκατομμύρια τσιγάρα ετησίω. Και επίσης ε, όλα υποστηρίζει πολλές από αυτέ τι δράσει κατάσχεση των κρατών μελών και είμαστε περήφανοι να αναφέρουμε ότι γύρω στα 500 εκατομμύρια τσιγάρα από αυτά που κατάσχουν τα κράτη-μέλη κατάσχονται ακριβώς με την υποστήριξη, με τη βοήθεια της όλα. Τώρα, ποιες είναι οι τάσεις που παρα, παρατηρούμε αυτή την περίοδο στο, ε, στην παράνομη αγορά. Ε, καταρχήν βλέπουμε μία τάση κατάσταση της παράνομης ε, παραγωγής αυτών των ε, προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε δηλαδή πλέον λαθρεμπόριο από τρίτες χώρες που εισέρχονται αυτά τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζουν και παρασκευάζονται εδώ, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να σας δώσω εδώ ένα-δύο παραδείγματα. Ε, πέρυσι, το Μάρτιο, ανακαλύφθηκε ένα εργοστάσιο σε μία από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και εκείνο που μας εξέπληξε ήταν ο όγκος της παραγωγής εκεί. Υπήρχαν 40 τόνοι καπνού που εντοπίστηκαν εκεί και η παραγωγική ικανότητα αυτού του παρανόμου εργοστασίου, αυτής της παράνομης παραγωγικής μονάδας ήταν 25 εκατομμύρια και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία ως προς ε, πώς είναι κατασκευασμένο τέτοιου είδους, ε, τέτοιου είδους μονάδες. Είδαμε, βρήκαμε 4,5 τόνους ε, ακατέργαστο καπνού, 7 εκατομμύρια τσιγάρα και 7 άτομα ε, κατασχέθηκαν και 7 άτομα με τέτοια υποσύλληψη. Και τώρα, μια δεύτερη τάση την οποία θα ήθελα να τονίσω είναι το γεγονός ότι δεν βλέπουμε μόνο ε, ε, τσιγάρα αλλά καπνό. Ε, που χρησιμοποιείται σε άλλες συσκευές καπνίσματος όπως λέει. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση ως έχει σήμερα σε ό,τι αφορά το παράνομο εμπόριο καπνού. Τι κάνουν τώρα ε, τα κράτη-μέλη και οι Ευρωπαϊκέ Αρχέ. Καταρχήν, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια πριν από γύρω στα 10 χρόνια και η πρώτη βασική πρωτοβουλία σε επίπεδο πολιτική ήταν ε, το σχέδιο δράση των Ανατολικών Συνόρων, γιατί είχαμε διαπιστώσει ακριβώ ότι τα Ανατολικά Σύνορα ήταν ιδιαίτερα ευάλωτα. Δύο χρόνια αργότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κατέρτισε ένα κείμενο στρατηγικέ ω προ το τι ακριβώ θα πρέπει να γίνει, με ποια μέσα θα πρέπει να επιτευχθούν όλα αυτά και επίση υπήρξε και ένα σχέδιο δράση που ακολούθησε και το οποίο εφαρμόστηκε για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ε, μετά λοιπόν ε, από την παρέλευση αυτών των ετών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπώνησε μια έκθεση προόδου όπου διαπιστώνει ότι παρά τις, ε, τα μέτρα που έχουν ληφθεί και την πρόοδο που έχουμε επιτύχει το πρόβλημα παραμένει γιατί αυτή η παράνομη δραστηριότητα είναι ακριβώς ε, ζημιογόνα και για την ε, δημόσια υγεία και για την, ε, τα δημόσια οικονομικά, τους δημόσιους πόρους αλλά και την ασφάλεια. Και γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα κατέληξε ένα δεύτερο σχέδιο δράσης που εστιάζει στους τομείς, τους ιδιαίτερα προβληματικούς στους οποίους έχουμε εντοπίσει. Η στρατηγική βέβαια του 2013 παραμένει επίκαιρη και σημαντική και επικαιροποιημένη και ε, όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, μόνο ο συνδυασμός της ε, σωστής επιβολής της νομοθεσίας μαζί με συντονισμένες δράσεις μπορούν να οδηγήσουν, οδηγήσουν στην καταπολέμηση, στην αποτελεσματική καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνού. Και αυτό που κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε είναι το να έχουμε ακριβώς ε, το κατάλληλο πλαίσιο και σε εσωτερικό και εξωτερικό πλαίσιο. Και ο κύριος τομέας πολιτικής τον οποίο εξετάζουμε είναι να είναι ασφαλής η διάβλη ε, του νόμιμου εμπορίου, ε, να κάνουμε τους σωστούς συνοριακούς ελέγχους ε, και να βελτιώσουμε τις ικανότητες εντοπισμού παρανόμου εμπορίου. Με βάση λοιπόν αυτές τις, αυτούς τους βασικούς άξονες, ποια είναι τα νέα στοιχεία που έχουμε συμπεριλάβει στο νέο σχέδιο δράσης. Έχουμε εντοπίσει λοιπόν τρει-τέσσερι τομεί οι οποίε έχουν προσθεθεί ω νέοι τομεί στο νέο σχέδιο δράση. Ε, καταρχήν, και αυτό μας γεμίζει με περηφάνεια, υπάρχει πλέον αυτή η σύμβαση ε, FCTC, το πρωτόκολλο ουσιαστικά της FCTC, μια δηλαδή σύμβαση η οποία έχει συναθρίσει υπό την αιγίδα και στα πλαίσια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και βέβαια έχουμε αναλάβει εδώ ηγετικό ρόλο σε Ευρωπαϊκή Ένωση και τέθηκε σε ισχύ το Δεκέμβριο του 2018 και έχουμε έξι χώρες εταίρους που έχουν προσπογράψει και έχουν κυρώσει αυτή την συμφωνία. Λοιπόν, αυτή, ε, αυτό το πρωτόκολλο της σύμβασης αποτελεί ε, τον, το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε τις προσπάθειες της ε, διεθνούς ανάληψης δράσης, αλλά ταυτόχρονα βέβαια συνεχίζουμε και τις προσπάθειες και σε διμερές επίπεδο. Επίσης, εξετάζουμε και στα στα, στα μέσα παραγωγής ε, για, την, για ε, για αυτά τα προϊόντα καπνού, γιατί βλέπουμε, όπω είπαμε, να υπάρχει μετεγκατάσταση τη ε, παραγωγή εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε προσπαθούμε να εστιάσουμε στα υλικά που χρησιμοποιούνται για την ε, παραγωγή. Και από εκεί και μετά, βέβαια, εξετάζουμε και τη μαύρη αγορά ω αγορά, την παράνομη αγορά. Δηλαδή, ω μια αγορά προσφορά και ζήτηση. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι αγοράζουν όλα αυτά τα προϊόντα καπνού, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα προσφέρονταν. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε περισσότερα έτσι ώστε να μειώσουμε τη ζήτηση για αυτά τα παράνομα προϊόντα καπνού ευαισθητοποιώντα περισσότερο το ευρύ κοινό. Ε, και εδώ συνεργαζόμαστε δηλαδή και με του συναδέλφου από τα ε, διάφορα τμήματα υγεία. Τώρα, να σας ε, αναφέρω τέσσερι, πέντε πιο συγκεκριμένε δράσει που περιλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο δράση, το οποίο γενικότερα περιλαμβάνει 50 στοιχεία, είτε αυτά έχουν να κάνουν με συμβάσει, είτε έχουν να κάνουν με εργαλεία πληροφορική, είτε με επιχειρησιακά θέματα. Καταρχήν, αναφέρθηκα στον κεντρικό ρόλο του πρωτοκόλλου FCTC γιατί υπήρχαν κάποιες ελλείψεις και τώρα έχουν πληρωθεί. Και βέβαια στο πλαίσιο της συνεργασίας με τρίτες χώρες ε, πάντα καλούμε αυτές τις χώρες να ε, υπογράψουν και να ε, κυρώσουν την, αυτό το πρωτόκολλο. Επίσης προσπαθούμε να γεφυρώσουμε χάσματα που υπήρχαν μέχρι τώρα στις διμερείς μας σχέσεις με γειτονικέ χώρες. Υπάρχει δηλαδή μια γειτονική χώρα με την οποία μέχρι τώρα δεν είχαμε την κατάλληλη ε, τελωνιακή συνεργασία. Πράγμα το οποίο εξετάζουμε αυτή την περίοδο ακριβώ για να δούμε αν μπορούμε να διορθώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση. Ένα τρίτο τώρα στοιχείο είναι το ότι θέλουμε να εξετάσουμε το τι θα κάνουμε με αυτά τα, τα μέσα ακριβώ ε, παραγωγή για την ε, παραγωγή προϊόντων εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, κυκλοφορούν νόμιμα τέτοιου είδου μηχανήματα, τέτοιου είδου εξοπλισμού εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, εξετάζουμε τα εργαλεία πληροφορική, τα οποία είναι πολύ σημαντικά σε ό,τι αφορά την τελωνιακή συνεργασία κατά του ε, συνορικού ελέγχου. Επίση, έχουμε και ένα ανεξάρτητο εργαστήριο προϊόντων καπνού, ε, στο οποίο γίνονται διάφοροι έλεγχοι των προϊόντων που κατάσχονται από τα κράτη-μέλη. Και επίση, δημιουργήσαμε και ένα ειδικό ευρωβαρόμετρο, το οποίο εξετάζει ακριβώ την ε, αντίληψη του ευρέω κοινού προ το τι ακριβώ θεωρεί σε σχέση με τα προϊόντα καπνού και το καθεξή. Και υπάρχουν και αξιωματικοί σύνδεσμοι ε, τη Όλαφ ε, ανά τον κόσμο. Εδώ δηλαδή σα έκανα μια πολύ δειγματοληπτική παρουσίαση των όσων έχουμε συμπεριλάβει στο σύνδεσμο σα και το τι κάνουμε, αλλά βέβαια είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Ευχαριστώ. Ωραία. Οι διαφάνειες αυτές θα δοθούν και στους ευρωβουλευτές. Ο κύριος Γκονζάλης πρώτα. Μια που το αίτημα απορρέει από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και μετά θα έχουμε καρστιά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση και πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπε η Όλαφ για το πρωτόκολλο αυτό, για τη σύμβαση πλαίσιο κυρίως, για τις κατασχήσεις μέσα ε, στο παράνομο αυτό εργοστάσιο, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπράβο που τα καταφέρατε. Έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πάντως συγχαρητήρια και για την βοήθεια του πρωτοκόλου. Ήδη το ότι υπάρχει αυτό το πρωτόκολλο το οποίο προβλέπει τον έλεγχο ε, παράνομων καπνών και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για καπνά που έρχονται απ' έξω είναι πολύ θετικό. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να συνειδητοποιήσει καλύτερα ε, την κατάσταση. Πρέπει δηλαδή να γνωρίζει ο κόσμος τι σημαίνει το να καταναλώνει κανείς παράνομα προϊόντα καπνού. Δεν μιλάω εδώ πέρα μόνο για τα καπνά που έχουν παραχθεί κυκλοφορούν νόμιμα και αυτά βέβαια κάνουν ζημιά, το ξέρουμε, ε, στην υγεία. Αλλά είναι και θέμα εδώ εσόδων, ε, διαφυγόντος κέρδους, όπως είπαμε. Ό,τι δουλειά γίνεται λοιπόν για να βρούμε και να καταπολεμήσουμε αυτά τα παράνομα προϊόντα καπνού είναι θετικό. Τώρα εγώ θα ήθελα να γνωρίζω αν έχετε εντοπίσει κάτι, γιατί ξέρετε τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένε Πολιτείες υπήρξε μεγάλη ανησυχία από τα ηλεκτρονικά ε, σιγαρέτα. Ξέρετε ότι ακόμα και νεκροί έχουν εντοπιστεί εξαιτίας του τσιγάρου αυτού. Και σίγουρα πολλοί έχουν ασθενήσει. Και έχει να κάνει αυτό μήπως και με παράνομα τέτοια τσιγάρα μήπως επειδή αναμειγνύονται και με άλλες ουσίες, με κανεβοειδή κλπ. Ή και άλλα ουσίες που δεν γνωρίζουμε, δηλαδή έχει εντοπιστεί καθόλου αυτή η δυνατότητα όπου εμπορευόμαστε τέτοια προϊόντα και μήπως και για μας μπορεί να είναι κάτι επικίνδυνο. Θέλω να το ξέρω. Πάντως σίγουρα πρέπει να εντοπίσουμε τα παράνομα προϊόντα και κάτι άλλο για το οποίο βέβαια δεν είναι υπεύθυνη η Όλαφ, να έχουμε την κατάλληλη νομοθεσία στο γενικότερο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Λοιπόν, θέλω να ξέρω αν εσείς από τη θέση σας, εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο αυτό, έχετε εντοπίσει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Άλλες ερωτήσεις παρακαλώ. από τα μέλη. 3, 2, 1, 0. Ωραία. Έκλεισε ο κατάλογος και επιστρέφουμε 5 λεπτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απαντήστε παρακαλώ στις ερωτήσει του κ. Γκονζάλης βέβαια πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ τον αξιότιμο Ευρωβουλευτή για τη στήριξή του και για τα καλά λόγια που είπε για το πρωτόκολλό μας. Συμφωνούμε και εμείς ότι αποτελεί στοιχείο κλειδί σε διεθνέ επίπεδο, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τον έλεγχο ε, προϊόντων καπνού. Προς το παρόν, όσον αφορά το φορολογικό, τα λαθρέα προϊόντα, τα σιγαρέτα, και το ξέρουμε εδώ και πολύ καιρό, ε, ισχύει αυτό το λαθρεμπόριο, βέβαια και για τα άλλα προϊόντα καπνού ε, που αναμειγνύονται με νερό. η φορολόγηση είναι μεγάλη και γι' αυτό το λαθρεμπόριο έχει προχωρήσει πολύ. Υπάρχουν και άλλα προϊόντα που δεν φορολογούνται τόσο πολύ και γι' αυτό ίσως κυρίως τα σιγαρέτα έχουμε ε, υψηλό λαθρεμπόριο. Δεν έχουμε λαθρεμπόριο δηλαδή στα άλλα προϊόντα ε, το ίδιο όσο και με τα κλασικά σιγαρέτα. Έχουμε και την κυρία Έμελιντ εδώ, μπορεί να πει ίσω περισσότερα για το θέμα των ελέγχων. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που μπορώ να σας πω για το ηλεκτρονικό τσιγάρο και για άλλες μορφές, όντως σε διάφορα σημεία του κόσμου έχουν αρχίσει κυβερνήσεις να αναλαμβάνουν δράση εμείς ποτέ δεν είπαμε ως Κομισιόν ότι είναι ασφαλή τα ηλεκτρονικά σιγαρέτα. Έχουν ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη οδηγίας ε, για τα καπνά, οπότε πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες που ακολουθούν και τα προϊόντα καπνών με ανώτατα επίπεδα νικοτίνης για παράδειγμα κλπ. Είναι δηλαδή ρυθμισμένα προϊόντα προς το παρόν. Και λέω προς το παρόν γιατί καμία χώρα μέλος δεν έχει αναφέρει τέτοιες περιπτώσεις, προβλήματα δηλαδή. Ρωτάμε, όπως επίσης κατά πόσο οι χώρες μέλη έχουν, πάρει κάποια, έχουν αναλάβει κάποια δράση, σκοπεύουν να αναλάβουν δράση. Όσον αφορά πάντως ένα από τα μεγάλα ζητήματα είναι τα αρωματικά, το οποίο είναι που αναμειγνύονται με τον καπνό, που είναι θέμα που είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Θα έπρεπε οι χώρες να τα απαγορεύσουν λοιπόν. Ωραία, ολοκληρώσαμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και σας ευχαριστούμε πολύ για το υλικό που προσφέρατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ακόμα και αν θα θέλαμε να είχαμε περισσότερους ευρωβουλευτές εδώ παρόντες. Λυπάμαι γι' αυτό. Πάντως να ξέρετε ότι εμείς θα στηρίξουμε τη δράση της Επιτροπής. Συνεπώς σας ευχαριστούμε πολύ. Αύριο το πρωί στις 9.30 αρχίζουμε. 9.30. 8.30 ε, είπε στην αρχή ο, ο πρόεδρος κατά λάθος. 9.30 αύριο λοιπόν.